68 μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 105 εδάφιο 6 του κανονισμού, εκφράστηκαν κατά τη σύσταση της Επιτροπής ΕΚΟΝ σε σχέση με την κατεξουσιοδότηση πράξης Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 114-49 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της 15ης ε, Μαΐου 2014 σε σχέση με τις ε, εισφορές για τους μηχανισμούς διεκπαιρέωσης. Και έτσι σε σχέση με αυτή τη σύσταση θα γίνει ψηφοφορία την Πέμπτη. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι σήμερα στις 5.17.00 και η προθεσμία για ξεχωριστές ή ονομαστικές ψηφοφορίες ή κατά τμήματα ψηφοφορίες. Η προθεσμία λήγει απόψε στις 19:07 η ώρα.